Καλωσορίζω την Επίτροπο κυρία Κράους και δίνω το λόγο στην εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν θα χρησιμοποιήσω τα τέσσερα λεπτά πιστεύω διότι τέτοια ώρα που είναι και τόσοι πολλοί που είμαστε δεν χρειάζεται να σας πω πολλά πράγματα. Ήθελα να πω ότι πρόκειται για μια έκθεση που αντιμετωπίζει ένα θέμα που τα επόμενα 10-15 χρόνια θα αλλάξει ριζικά τη σχέση μεταξύ ατόμων και πραγμάτων και μεταξύ πραγμάτων και πραγμάτων. Μια νέα εφαρμογή του ίντερνετ είναι. Θέλω να συγχαρώ εδώ την Επιτροπή για την ανακοίνωση που παρουσίασε, διότι είναι σκόπιμη αυτή την ώρα. Πρόκειται για ένα μας επιτρέπει να μπορέσουμε να προβλέψουμε τις συνέπειες αυτής της νέας εφαρμογής. Συνέπειες που έχουν πολλά θετικά, μπορεί να βελτιώσουν πολλά κομμάτια της ζωής μας, ανοίγουν ε, ε, δυνατότητες νέων ε, δραστηριοτήτων, βελτίωση της παραγωγής, αλλά περιλαμβάνουν και κινδύνους. Προφανώς και η έκθεση που επεξεργάστηκα μαζί με τους και συγητές των άλλων πολιτικών ομάδων, με τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω για τη δουλειά τους, προσπαθήσαμε να επιτρέψουμε στους χρήστες να έχουν όλη την εξασφάλιση και την ιδιωτική και τη δυνατότητα, ιδιωτική δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις νέες αυτές τεχνολογίες. Ε, μελετήσαμε για να δούμε κατά πόσον όλο αυτό το πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο, κάλυπτε τις δυνατότητες, όλες τις δυνατότητες που θα υπήρχαν ε, με τις νέες εφαρμογές από ό,τι φαίνεται προς το παρόν τούτο συμβαίνει. Αυτό που συμφωνήσαμε ωστόσο είναι όσο ενσωματώνονται οι εφαρμογές αυτές τις διάφορες διαστάσεις της ζωής μας να προχωρούμε σε αξιολόγηση επιτόπου ώστε να ξέρουμε ότι υπάρχει κάλυψη της ιδιωτικής ζωής των χρηστών και της ασφάλειάς τους και από την υγεία και την προσωπική ζωή και μια σειρά άλλων ζητημάτων. Είναι μια σωστή έμφαση αυτή που δίνουμε. Το ξεκίνημα είναι πέραν αυτών που αναφέρει η έκθεση, θα ήθελα να προσθέσω, κυρία Επίτροπε, το ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ενημερώσουμε σωστά τους χρήστες, ώστε να γνωρίζουν πραγματικά περί τίνος πρόκειται. Διότι στην πραγματικότητα λέμε χρήστες, αλλά αν μιλήσετε με τους περισσότερους βουλευτές στο σώμα που δεν ασχολούνται με τέτοια ζητήματα, θα διαπιστώσετε ότι όταν τους λέμε ίντερνετ των πραγμάτων μας κοιτάνε ε, με γουρλωμένα μάτια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον, πέραν όλων αυτών των δυνατοτήτων και των στοιχείων που περιλαμβάνει η έκθεση και η ανακοίνωσή να σκεφτούμε καλύτερα πώς θα εξηγήσουμε στον κόσμο, στους πολίτες, στους χρήστες, τι σημαίνει η ίντερνετ των πραγμάτων. Και τι μπορεί να δημιουργηθεί με τις νέες αυτές εφαρμογές και πώς καλύπτονται η προσωπική του ζωή, η ασφάλειά τους. Αυτό είναι το κεντρικό στοιχείο της νέας εφαρμογής. Να εμπιστευθούν αυτό το νέο σύστημα οι πολίτες. Τίποτα άλλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω πολλούς ομιλητές για αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν η κυρία Κολόνσκα Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Το ίντερνετ των πραγμάτων είναι κομμάτι της ε, ψηφιακής ε, ατζέντα ε, και στόχος της βεβαίως είναι η πρόσβαση στο ίντερνετ παντού πρέπει να παλέψουμε επίσης την, ε, τον ψηφιακό αποκλεισμό στη χώρα μου παραδείγματος χάρη μόνο 13% των οικογενειών έχουν ευρυζωνική σύνδεση. Προτείνεται λοιπόν πως μέχρι το 2013 θα πρέπει να υπάρχει γενική πρόσβαση στο ίντερνετ. Αυτό είναι σωστό. Μιλάμε τώρα για ένα ίντερνετ των πραγμάτων. Μιλάμε για πράγματα τα οποία εντωμεταξύ ήδη υπάρχουν. Και ελπίζουμε να μην γίνει ακόμη μεγαλύτερη η ψαλίδα. Γιατί φοβόμαστε πως θα οδηγηθούμε σε ένα νέο κύμα ψηφιακού αποκλεισμού στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτοί οι οποίοι μαθαίνουν το ίντερνετ ε, τώρα ε, να έχουν μικρότερη γνώση από αυτούς που το γνώριζαν εδώ και χρόνια θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και να το δει η Κομισιόν για να μην δημιουργηθούν αυτές οι διαφορές τις οποίες ανέφερα. Σας ευχαριστώ η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η οικονομική ανάκαμψη σημαίνει πως χρειαζόμαστε την τεχνολογία και έτσι θα οδηγηθούμε στην ανάπτυξη. Το ίντερνετ των πραγμάτων θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ανάγκες αναπήρων, ηλικιωμένων, αλλά θα πρέπει βεβαίως να προστατεύσουμε την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων, να είναι εύκολη η πρόσβαση και να ενημερώσουμε τους πελάτες για το τι υπάρχει από πλευράς υπηρεσιών. Πρέπει η Κομισιόν λοιπόν να εφαρμόσει τους κανονισμούς που ήδη υπάρχουν και να παρουσιάσει ένα χρονοδιάγραμμα για τις ε, κατευθυντήριες γραμμές που θέλει να προτείνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο RFID. Θα πρέπει επίσης αυτό να συνοδευτεί από μέτρα όπως το να μην υπάρχει ανιχνευσιμότητα του IP της διεύθυνσης αυτής. Νικολάου. Νικολάου. για την πολύ καλή εργασία της. Πράγματι, αυτή η συζήτηση αναφέρεται στο μέλλον και αναφερόμαστε σε μια επανάσταση κατά κάποιο τρόπο στην επικοινωνία, στην επικοινωνία ανθρώπων και πραγμάτων αλλά και συσκευών μεταξύ τους. Και παράλληλα με την πρόκληση που έχει αυτή η συζήτηση και είναι προς τιμή νομίζω του Κοινοβουλίου μας ότι έχουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα και όλες αυτές τις δράσεις και την έκθεση αυτή ε, πρέπει να δούμε και του κινδύνου που αυτή ελοχεύει καθώ χρησιμοποιεί τεχνολογίε αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων οι οποίε περιέχουν πρόσβαση στην ιδιωτική ζωή και ο κίνδυνο που ανακύπτει είναι σαφή πρόσβαση και προστασία αλλά και ευρυζωνικότητα από τη μία σε αντιπαράθεση με την ιδιωτικότητα. οι προβληματισμοί είναι εμφανεί ποιο θα τη διοικεί τι θα γίνει με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πόσο ιδιωτικά θα είναι τελικά αυτά τα δεδομένα μας πόσο καλή ασφάλεια θα υπάρξει. αυτό που χρειάζεται είναι η ισορροπία στη νέα αυτή τεχνολογία μια τεχνολογία η οποία θα πρέπει να είναι αξιόπιστη μια τεχνολογία η οποία στην επεξεργασία των δεδομένων θα σέβεται απολύτως τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρόιτευα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Για κάποια, για αρκετά χρόνια βλέπουμε πως το ίντερνετ αλλάζει τον κόσμο μας ριζικά μερικές φορές και νομίζω ότι βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της ψηφιακής επανάστασης. Μου άρεσε η έκθεση της κυρίας Μπαντερικούσετ διότι τονίζει την ανάγκη νέας νομοθεσίας στον τομέα την ανάγκη υποστήριξης επιπλέον υποδομών για το ίντερνετ και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Τέλος, πρέπει να μπορούμε να προεξοφλούμε τους κινδύνους για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου. Χρειάζεται πάντα μια γρήγορη, σωστή αξιολόγηση των συνεπειών των ραδιοσυχνοτήτων και οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν τη συνέχεια, τη, επίπτωση κάθε ε, δεδομένο έχει στην ζωή τους. Θα πρέπει να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στους πολίτες μας να ζουν και να χρησιμοποιούν τα τσίπ αυτά με ασφαλή τρόπο, αλλά να μην υπάρχουν καταχρήσεις. Και ταυτόχρονα πρέπει να, να δώσουμε και ένα σαφές μήνυμα προς την Κομισιόν. Ο κύριος Πασκά τελευταίος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να υποστηρίξω αυτή την έκθεση η οποία πράγματι ανοίγει το δρόμο για την εισαγωγή μελλοντικής τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας. Πρόκειται για τεχνολογίες ε, οι οποίες θα δώσουν νέα πνοή στην ανάπτυξη και θα αλλάξουν τη ζωή των πολιτών μας. Είναι τεχνολογίες που θα εισαγάγουν νέα στοιχεία στις υπηρεσίες και στα προϊόντα. Σε σχέση όμως με αυτές τις νέες τεχνολογίες όμως πρέπει σοβαρά να εξετάσουμε πώς θα έχουμε νομική διασφάλιση της ιδιωτική ζωής των πολιτών. Διότι αυτές οι νέες τεχνολογίες θα παρακολουθούν, θα ειχνηλατούν, όχι μόνο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αλλά και τους χρήστες τους. Συνεπώς από τη στιγμή που θα λειτουργεί αυτή η τεχνολογία δεν πρέπει να παραβιάζει την ιδιωτική ζωή. Ευχαριστώ. Δίνω τώρα το λόγο στην Επίτροπο Κρός εκ μέρους της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με μεγάλο θαυμασμό για την κυρία Μπάντια Ικούτσια θα προσπαθήσω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο. Και πράγματι το Ευρωκοινοβούλιο υπήρξε ενεργό και συμμετείχε σημαντικά και σφαιρικά θα έλεγα στην προώθηση των θεμάτων διαδικτύου. Πρέπει να σας πω στην έκθεσή σας διατυπώνεται πολύ σωστά την ανάγκη παρακολούθησης των νέων εξελίξεων που θα επηρεάσουν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών στις μεταγενέστερες δεκαετίες. Με εντυπωσίασαν επίσης οι ομιλίες των βουλευτών που επένεσαν το έργο της κυρίας Συμπάντια και με, ε, με συγκίνησε το ενδιαφέρον που δείξατε για τους πολίτες. Είναι και θέμα επικοινωνίας βεβαίως, διότι θα πρέπει να αποδώσουμε περισσότερη προσοχή σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Συγχαίρω λοιπόν τον πρωτοπόρο σας ρόλο στην υπογράμμιση των μεταβολο... κρίσιμων μεταβολών στο διαδίκτυο και πρέπει να πω ότι πραγματικά η συγκήτρια έκανε θαυμάσιο θαυμάσια δουλειά υπογραμμίζοντας τα δημόσια θέματα. Και συμφωνώ ότι πρέπει να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο. Πρόσφατα μίλησα για το πλαίσιο αξιών που πρέπει να προστατεύσουν τον Ευρωπαίο πολίτη προωθώντας ταυτόχρονα τις επενδύσεις στον κρατικό και στον ιδιωτικό τομέα για το διαδίκτυο των πραγμάτων. Για να αναπτυχθεί λοιπόν αυτό το διαδίκτυο των πραγμάτων αποτελεσματικά, χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα να έχουμε μια ευρεία δημόσια συζήτηση, να εξασφαλίσουμε σταθερούς όρους επενδύσεων και σίγουρα πρέπει να αποφύγουμε οι πολίτες να αισθάνονται ότι το διαδίκτυο των πραγμάτων τους επιβλήθη Υποχρεωτικά δηλαδή. Δεν υπάρχει τέτοια υποχρεωτικότητα. Το θέμα είναι να δώσουμε, να απαντήσουμε στην πρόκληση και να δώσουμε μια ευκαιρία και οι τα ενδεχόμενα αποτελέσματα μπορεί να, είναι, να μεγαλουργήσουν. Πρέπει να έχουμε συνείδηση όμως των βημάτων που ε, ε, πραγματοποιούμε και πρέπει να εξασφαλίσουμε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνθήκες επενδύσεων μαζί με κοινού κανόνες. Είναι μια πρόκληση που και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν στο οποίο πρέπει να ανταποκριθούμε. Τώρα λοιπόν που έχουμε μια ατζέντα ήρθε η ώρα για να κάνουμε την πραγματική δουλειά και να αρχίσουμε να περάσουμε στην εφαρμογή. Πράγματι έχουμε ξεκινήσει να ακολουθούμε το δρόμο τώρα όμως θα πρέπει να περάσουμε στην εφαρμογή και από τις 14 ε, ε, τα 14 θέματα που περιλάβαμε στην ανακοίνωσή μας πρέπει να σας πω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Η, μια μελέτη όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ραδιοσυγνωτήτων ε, προχωρεί και ο διαθεσμικός διάλογος επίσης. Πιο μακρόπνοα πρέπει να σας πω ότι ένα πρώτο κύμα, κύμα 8 ε, ερευνών με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ολοκληρωθεί φέτος και θα μελετήσουμε τις συνεργίες του μέλλοντος. Υπάρχουν και άλλες δράσεις, διακυβέρνηση του διαδικτύου, η απόφαση για τη σίγαση ε, η ιδιωτική ζωή και η προστασία των ιδιωτικών δεδομένων. Χρειάζεται δέσμευση και συλλογική προσπάθεια για να τα πετύχουμε. Γι' αυτό, κυρία Πρόεδρε, αποφάσισα να συστήσω μια ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα ανασκοπήσει αυτά τα θέματα μεταξύ άλλων και θα συντίθεται από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, του κλάδου, των πανεπιστήμιων, των κυβερνήσεων και θα συναντούνται κάθε τρίμηνο για δύο χρόνια και βεβαίως θα μας αναφέρουν σχετικά με την πρόοδό τους και όλα αυτά θα είναι στη διάθεσή σας. Καταλήγοντας θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά έχουν σχέση με την επικοινωνία και πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί στους λαούς. Θα ήθελα ένα σχόλιο ακόμη να κάνω. Πράγματι, είναι σαφές ότι η Κομισιό έχει κάνει τη δήλωση ότι θα έπρεπε κάθε Ευρωπαίος να είναι ψηφιακός το 2013. Το πιστεύουμε αυτό. Και όχι μόνο το πιστεύουμε, αλλά θα το πράξουμε και μπορούμε να το πράξουμε. Και έχω το προνόμιο να ε, καλέσω την ε, Επιτροπή Ήτρα και την Επιτροπή Πολιτισμού Και υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία έχουμε περιλάβει σε ένα κατάλογο πράξεων που πρέπει να προχωρήσουν. Κάθε Ευρωπαίος πρέπει να γίνει ψηφιακός και ελπίζω ότι με αυτόν τον τρόπο καλύπτω την ανησυχία σας. Προστασία λοιπόν των προσωπικών δεδομένων. Είναι και πολύ σημαντικό, και αυτό στην ατζέντα μας. Είναι θέμα εμπιστοσύνη και ασφάλειας. Εάν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν μπορεί να αναμένεται οι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν αυτό το φαινόμενο, αν μπορώ να το αποκαλέσω έτσι. Δηλαδή είναι ένας κύκλος που, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για να είναι η πρόκληση ικανοποιητική για τον Ευρωπαίο πολίτη. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Έληξε συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Και τώρα περνάμε στο επόμενο μας θέμα. Η σημερινή διάταξης τη διακυβέρνηση του διαδικτύου έκθεση του κυρίου Σώσα Βάγνερ